είναι η ενίσχυση της καινοτομίας και της οικονομικής ανάπτυξης στο πλαίσιο της μελλοντική ευρωπαϊκής διαχείρισης γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Θα δώσω το λόγο στον εισηγητή, τον κύριο Χάουτεμα. Τέσσερα λεπτά παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, κύριε Επίτροπε, έχουμε μιλήσει για διάφορα προβλήματα, αλλά μία από τις αιτήσει είναι η ίδια η πολιτική. Υπάρχουν τεράστιες ευκαιρίες για τους γεωργούς σήμερα και είναι δικιά μας ευθύνη να δώσουμε τα περιθώρια, την ευκαιρία αυτή που έχουν οι γεωργοί να την αρπάξουν και να έχουν αποτελέσματα. Βρίσκομαι εδώ και είμαι ευγνώμων προς τους συναδέλφους στην Επιτροπή Γεωργίας που με βοήθησαν να εκπονήσω την έκθεση αυτή. Πολλά αλλάζουν και αυτό πρέπει να το έχουμε υπόψη μας και πρέπει να φροντίσουμε να υπάρχει και μεγαλύτερη αντίσταση στα παράσιτα των καλλιεργιών μας. Γι' αυτό και χρειαζόμαστε την καινοτομία. Η πρόκληση είναι μεγάλη. Χρειάζεται γνώση, καινοτομία που μπορεί να βοηθήσει να έχουμε καλύτερα τρόφιμα και αρκετά και συγχρόνως να προστατεύουμε το περιβάλλον και να βελτιώσουμε την ποικιλία. Είμαι περήφανος λοιπόν για το αποτέλεσμα. Η παλιά νομοθεσία παροχημένη πρέπει να αλλάξει, να αντικατασταθεί να υπάρχει έλεγχο των καλλιεργών μας, να χρησιμοποιούμε τις καλύτερες δυνατόν πρακτικές για όλα μας τα προϊόντα, για τα λοιπάσματα κλπ. Θεωρώ ότι είναι χρέος μου να βοηθήσω τους γεωργούς ότι οι κακοί και παροχημένοι πρακτική ακολουθούν να την εγκαταλείψουν και να φροντίσουν για την προστασία του περιβάλλοντος. Αυτό θα γίνει άμα δώσουμε περιθώριο στους γεωργούς για να τα καταφέρουν και αυτό είναι το κύριο μήνυμα χώρος για καινοτομία, επιχειρηματικότητα στη Γεωργία. Οι δυνατότητες που έχει ο τομέας είναι τεράστιες. Με την κατάλληλη ρύθμιση που να μην είναι εμπόδιο, θα μπορέσουν οι Γεωργοί να αποφεληθούν πλήρως από τις νέες ευκαιρίες. Πρέπει να τους δώσουμε λοιπόν περιθώριο και να μην περιορίσουμε τις δυνατότητές τους. Κανείς δεν γνωρίζει καλύτερα τη δουλειά τους από τους ίδιους τους γεωργούς. Ας τους αφήσουμε λοιπόν μόνοι τους να αποφασίσουμε πώς, με, ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος για να πετύχουν τους στόχους τους. Πρέπει να τους δώσουμε περιθώρια για νέες ιδέες και καινοτομία. Να μην τους δώσουμε ένα checklist, ένα κατάλογο δηλαδή εμείς που καθόμαστε πίσω από τα γραφεία μας. Νέοι κανόνες λοιπόν, οι οποίοι θα αποφέρουν κέρδη στο μέλλον νέες ε, εφαρμογές να δοκιμαστούν. Η Γεωργία έχει τη δυνατότητα να προσφέρει στην αυριανή οικονομία εφόσον χρησιμοποιήσουμε καλά τις δυνάμεις της φύσης θα ενισχύσουμε την οικονομία μας. Να χρησιμοποιήσουμε φυσικά μέσα για την παραγωγή έτσι και οι καταναλωτές θα εξυπηρετηθούν καλύτερα αλλά και θα περιορίσουμε τις εκπομπές του οξυδίου του άνθρακα. Έτσι λοιπόν, η αυριανή γεωργία πρέπει να το ξέρουν όλοι, έχει φτάσει. Αρκεί να τους το επιτρέψουμε και η πολιτική αλλά και ο κλάδος. Η έκθεσή μου λοιπόν προσφέρει νέες δυνατότητες. Ελπίζω αύριο όλοι οι συνάδελφοι να με υποστηρίξουν στην έκκλησή μου για να βοηθήσουμε τους γεωργούς να μας προσφέρουν τη γεωργία του μέλλοντος. Πραγματογνωμοσύνη από τους ίδιους τους γεωργούς χρειάζεται. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρος. Ευχαριστώ. Έχουμε... Επτά μέλη τα οποία ζήτησαν τον λόγο. Θα δώσουμε το χρόνο σε όλους και ξεκινάμε με την κυρία Πέτυρ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Μία απαιτητική κοινή αγροτική πολιτική και επιτυχημένη και εγγύηση προϊόντος ποιότητας, ε, όλα αυτά είναι τότε από την εξέλιξη της γεωργίας και της απαραίτητης ε, χρηματοδότησης σε όλα τα επίπεδα. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να έχουμε βιώσιμες ε, περιοχές της υπαίθρου και βιώσιμο εμπόριο και κατανάλωση. Ο εισηγητής αποδέχτηκε τις τροπολογίες μου και έτσι έδωσε τη δέουσα σημασία στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες σίγουρα συνεισφέρουν στην ανάπτυξη των περιοχών της υπαίθρου και στην προστασία του, της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς. Πρέπει να δούμε τη γεωργία με άλλο πνεύμα, σε ε, συγκεκριμένο επίπεδο το οποίο θα απευθύνεται στους καταναλωτές και αναγνωρίζοντας και την προστιθέμενη αξία της γεωργίας σε όλο τον κόσμο. Εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να παραμείνει το θέμα το οποίο σχετίζεται ε, στους καταναλωτές και θα βασίζεται στην τεχνολογία και στις ε, γνώσεις. Ο κύριος Σερανόζα. Η καινοτομία στη γεωργία απαιτεί σημαντική επένδυση στην έρευνα και την ανάπτυξη και την υποστήριξη των γεωργών για να βρουν τις κατάλληλες λύσεις καινοτόμες μορφές γεωργίας όπως αυτή η οποία είναι η γεωργία ακρίβειας θα πρέπει να έχουν μια σωστή σχέση κόστους ωφέλους και να δίνουν τις δυνατότητες για τις πιο μικρές αγροτικές ε, εκμεταλλεύσεις όπως αυτές που βρίσκονται σε υπερπεριφερειακές ή απομονωμένες περιοχές να λειτουργήσουν ιδίω στις περιοχές που η γεωργία είναι απαραίτητη για την τοπική οικονομία. Θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε λοιπόν με τον τρόπο αυτό την ε, πρόκληση της κλιματικής αλλαγής. Γι' αυτό είναι απαραίτητο να χρησιμοποιήσουμε κάθε τεχνολογία που δίνει καινοτόμε λύσεις με διαφορετική χρήση των πρακτικών. Θα πρέπει όμως για να γίνει αυτό η γεωργία να είναι στο κέντρο της προσοχής μας να είναι η κύριη ε, αλλαγής και θα πρέπει να τύχουν τις πλήρους προσοχής μας. Ευχαριστώ. Ουσιακών και βιολογικών καλλιεργειών είναι η καλύτερη, ίσως και η μοναδική απάντηση στο αμερικανικό μοντέλο γεωργίας το μαρικανικό μοντέλο αυτό που κάποιοι και μέσα στην ευρώπη επιχειρούν να μας επιβάλλουν μέσω της ttip. είναι σίγουρα πολύ αποτελεσματικό μόνο για τους κολοσσούς του αγροτοδιατροφικού τομέα και τα λόμπι των μεγάλων παραγωγών. είναι όμως καταστροφικό για το περιβάλλον την υγεία μας τις μελλοντικές γενιές. είναι καταστροφικό και για τα είκοσι εκατομμύρια αγρότες των χωρών της ευρώπης που στην πλειοψηφία τους επέλεξαν και κατάφεραν με σκληρούς αγώνες να διατηρήσουν μια άλλη οργάνωση της παραγωγής αντί λοιπόν να τραβάει το χαλί κάτω από τα πόδια του η ευρωπαϊκή ένωση πρέπει να στηρίξει αυτή την κληρονομιά. δεν υπάρχει κανένα καλό συμβιβασμό για την ttip. το ευρωπαϊκό μοντέλο παραγωγή στηριγμένο στη μικρή μονάδα βρίσκεται στον αντίποδα αυτού που ζητούν οι αμερικανικέ και ευρωπαϊκέ πολυεθνικέ. σε μια εποχή που η βιωσιμότητα έχει καταστεί ζητούμενο και η δέσμευση των περισσότερων μεγάλων οικονομιών του πλανήτη υπάρχει η καταστροφή του ευρωπαϊκού παραγωγικού ιστού θα αποτελέσει

Ευχαριστώ. Η καινοτομία εξακολουθεί να αποτελεί προτεραιότητα για την ε, γεωργία σήμερα, δεδομένου ότι έχουμε κλιματική αλλαγή, αυξάνεται η ζήτηση σε τρόφιμα και υπάρχουν και απειλέ ε, για το κλίμα. Πρέπει να υποστηρίξουμε λοιπόν τη γεωργία ώστε να μπορέσουμε να αυξήσουμε την παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα του τομέα. Με άλλα λόγια, οι αγρότες θα χρειαστεί να παράγουν περισσότερα με λιγότερα στο μέλλον. Ωστόσο, η προσαρμογή των νέων τεχνολογιών της γεωργίας από τους Ευρωπαίους αγρότες μέχρι τώρα έχει γίνει με πολύ διλαβήματα. Η πρόκληση λοιπόν κύριε Επίτροπε είναι να υποστηρίξουμε την ε, μεταφορά γνώσης από τους ερευνητές τους γεωργούς με χρήση καινοτόμων τεχνικών που επικαιροποιούν τη σχετική νομοθεσία καθώς επίσης και την ε, δημιουργία κατάλληλων δυνατοτήτων χρηματοδότησης για τους γεωργούς. Πολλές από τις εκμεταλλεύσεις σήμερα δεν έχουν σχέση με τις ε, εκμεταλλεύσεις της δεκαετίας του 50. Και αν τα καταφέρουμε, οι γεωργοί του 2050 μάλλον θα διαφέρουν πολύ ε, από τους γεωργούς του σήμερα. Ευχαριστώ πολύ. Επόμενος ομιλητής, ο κύριος Σεμπαστιά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε συζητούμε κάτι πάρα πολύ σημαντικό για τη γεωργία, όπω είναι η καινοτομία. Σίγουρα πρόκειται για ένα ακόμα στοιχείο, αλλά όχι το μόνο Πρέπει να ξεφύγει από την κρίση που έχει, ε, στην οποία έχει περιέλθει ο τομέα. Και ε, ε, αυτό και συζητούμε τα μέτρα τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η καινοτομία μπορεί να έχει διάφορε πτυχέ και γι' αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή, ο οποίο διευκρίνησε ότι η καινοτομία και βιωσιμότητα δεν είναι απομακρυσμένα. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε μια γεωργία που δεν θα εξαρτάται από αγροχημικά προϊόντα και θα μπορέσουμε να έχουμε φθηνότερη παραγωγή προϊόντων και να μπορέσουμε ταυτόχρονα και να προστατεύουμε τη βιοποικιλότητα. Το να έχουμε βιώσιμη γεωργία σημαίνει ότι δεν θα πρέπει να παραμείνουμε στο παρελθόν, θα πρέπει να κοιτάμε το μέλλον και να προσπαθήσουμε να έχουμε μια αποτελεσματική και διαρκή γεωργία με μια ασφαλή και μόνιμη διαδικασία. Ίσως το πιο καινοτόμο στοιχείο θα είναι να εκμεταλλευτούμε όλη τη δύναμη που μας προσφέρει η φύση και την οποία έχουμε ξεχάσει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Σύμφωνο ότι οι καινοτόμε τεχνικές στην γεωργία είναι πολύ σημαντικές και πρέπει να έχουμε και πιο επίκαιρη πληροφόρηση από την Κομισιόν για να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε ότι η κοινή γνώμη θα υποστηρίξει αυτό το εγχείρημα και δεν θα καταφερθεί εναντίον του. Θα πρέπει να έχουμε καλύτερη σύνδεση μεταξύ έρευνας και εφαρμογής Είχαμε πρόσφατα τη συζήτηση για τον γλυφοσάτ στην, ε, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ένα από τα θέματα τα οποία μας ενδιαφέρουν ακριβώς πώς θα, θα αντικαταστήσουμε τα προηγούμενα παραστοκτόνα. Αλλά οι γεωργοί δεν γνωρίζουν όλες αυτές τις λεπτομέρειες. Για όλο αυτό το λόγο η Κομισιόν θα πρέπει να δίνει μεγαλύτερη σημασία στην χρήση της καινοτομίας στην γεωργία. Κύριος Καπούτο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε αποτελεσματική και καινοτόμως γεωργία ε, μας χρειάζεται για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τις προσκλήσεις της βιωσιμότητες που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι μικρές εκμεταλλεύσεις. Η σύγχρονη αγροτική εκμετάλλευση δεν σχετίζεται μόνο με την παραγωγή αγαθών, αλλά πρέπει να λειτουργήσει σε πολλέ ε, πτυχέ. Θα πρέπει να κάνει μεταποίηση προϊόντων, άμεση πώληση και αγροτουρισμό βασίζονται στην τεχνολογία της πληροφορικής και της επικοινωνίας ε, βάση παρακολούθησης στοιχείων σε πραγματικό χρόνο, τεχνολογίες αισθητήρων και συστήματα καινοτομία για τη βελτιστοποίηση των συστημάτων παραγωγής ή της ε, γεωργίας ακριβίας. Όλα αυτά θα μας επιτρέψουν να έχουμε καλύτερο έλεγχο ε, και καλύτερη παρακολούθηση των καλλιεργειών. Πιστεύω ότι οι σύγχρονες τεχνολογίες θα μας βοηθήσουν να κάνουμε πιο δελαστική τη γεωργία για τους νέους αγρότες και γι' αυτό ακριβώ ε, θεωρώ ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να κάνει περισσότερα ώστε να ευνοήσει την καινοτομία στη γεωργία. Ευχαριστώ πολύ. Με αυτό ολοκληρώνεται η διαδικασία του ΚΑΤΣΙΑΗ. Να δώσω τώρα το λόγο στον Επίτροπο. Επίτροπε Χόγκαν, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Χατωμά, τον εισηγητή, για την εκπόνηση και την παρουσίαση τη έκθεση αυτή όσον αφορά την ενίσχυση τη καινοτομία και τη οικονομική ανάπτυξη στα πλαίσια τη μελλοντική ευρωπαϊκή διαχείριση. Από τι συζητήσει που είχα μαζί του, ξέρω πόσο πολύ ενδιαφέρεται για αυτά τα θέματα. Και εγώ στηρίζω τα όσα λέει. Οι προκλήσει είναι πολύ σημαντικέ που αντιμετωπίζει ο κλάδο. Γιατί η καινοτομία είναι τόσο σημαντική. Η καινοτομία επιτρέπει στον κλάδο να αναπτύξει νέα προϊόντα, νέες μεθόδους, υπηρεσίες και να ανταποκριθεί σε προκλήσεις όπως είναι κλιματική αλλαγή, αλλά και άλλες κοινωνικές ακόμα προκλήσεις, αλλά και περιβαλλοντικές, αλλά και άλλες όπως είναι ανταγωνιστικότητα. Όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι πρέπει να υπάρξει διάθεση επαρκής τροφίμων, άρα χρειαζόμαστε μια καλύτερη παραγωγή, πιο βιώσιμη. Πολύ σωστά Εκπώνησε λοιπόν την έκθεσή του και οι προτάσεις του κύριου Χέτεμα είναι σωστές. Ε, ζητάει διάφορες δράσεις από πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που τις παίρνουμε πολύ σωστά υπόψη. Την χρήση της τεχνολογίας, τα αντιμικροβιακά ε, φάρμακα. Για όλη την καινοτομία η Επιτροπή θα δράσει. Η επικουρικότητα όμως πρέπει πάντα να λαμβάνεται υπόψη. Τοπικά προβλήματα απαιτούν τοπικές λύσεις και η Επιτροπή δεν είναι η καλύτερη σε θέση πάντα να προτείνει λύσεις. Μερικές φορές οι λύσεις πρέπει να βρεθούν σε περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο. Πάντως σίγουρα χρειάζεται να προσπαθήσουμε να έχουμε νέες πρακτικές, νέες μεθόδους. Αυτό σημαίνει καινοτομία. Και θα ήταν καλό να επενθυμίσω πόσο στο τωρινό πολιτικό μείγμα, policy mix, Μίγμα πολιτικής χρησιμοποιούμε την καινοτομία. Τη στηρίζουμε με τον Horizon 2020 που είναι για την έρευνα και την καινοτομία. Για τη δασοκομεία επίσης και εκεί στηρίζουμε την καινοτομία. Κοινωνικές προκλήσεις, ε, ε ασφαλής διάθεση τροφίμων, έρευνα ε, στο θαλάσσιο περιβάλλον, στα εσωτερικά ύδατα. Για το 2016 και 2017 έχουμε διάφορα προγράμματα. Στα πλαίσια του Horizon 2020 θα δείτε ότι αντιμετωπίζουμε πολλά από τα προβλήματα που αναφέρονται στην έκθεση. Το πρόγραμμα εργασίας για το 2016 και 2017 δείχνει ότι το Horizon 2020 είναι ε, το μεγαλύτερο πρόγραμμα, περισσότερο πρικοδοτημένο από οποιοδήποτε άλλο ποτέ. Η διαχείριση όμως γίνεται και από τη Γενική Διεύθυνση Άκρη και από τη Γενική Διεύθυνση για την έρευνα. Για αυτά χρόνια έχουμε με πέντε δις το νορίζοντα 2020. 71 θέματα από τη Γεωργία. 671 εκατομμύρια χρηματοδότηση για πάρα πολλά προγράμματα, 14 ξεκίνησαν ήδη το 2014, 22 θα αρχίσουν τώρα και άλλα θα υποβληθούν στη συνέχεια. Τα τελευταία τρία χρόνια, 2017 δηλαδή μέχρι 2020, θα ξέρουμε το Σεπτέμβριο του 2017 ακριβώς τι θα καλύψει. 94 προγράμματα πάντως έχουν να κάνουν με την πρόσφατη προγραμματική περίοδο. Προγράμματα θα εφαρμοστούν σε 24 χώρες. Ξέρω ότι μερικές φορές ακούγεται ότι είναι κατακαιρματισμένη η εφαρμογή του οράζο 2020. Όμως υπάρχει επικουρικότητα. Και μόνο με την επικουρικότητα μπορούμε να φτάσουμε σε ολόκληρη την Ευρώπη με τον κατάλληλο τρόπο. Πιστεύουμε ότι το μείγμα πολιτικής μας είναι το σωστό. Φυσικά πρέπει να κοιτάμε επικριτικά τα διάφορα μέσα χρηματοδότησης που έχουμε για να δούμε μήπως μπορούμε να τα βελτιώσουμε. Στην άτυπη συνάντηση των Υπουργών ε, Γεωργίας ε, πήγα στην χώρα του κύριου Χάιτεμα και εκεί επισκεφτήκαμε και την έκθεση τροφίμων η οποία ήταν ακριβώς αφιερωμένη στην καινοτομία στα τρόφιμα και εκεί είδαμε ε, χρήση καινοτόμα της τεχνολογίας που πραγματικά μας ενθουσίασε. Όλοι εντυπωσιαστήκαμε από αυτά που είδαμε γιατί δείχνουν ακριβώς όλα αυτά τα ζητήματα τα οποία σας απασχολούν και αναφέρατε και εσείς σήμερα εδώ στη συζήτηση. Η ανάπτυξη της τεχνολογίας, οι επενδύσεις και πώς αυτή θα χρησιμοποιηθεί στην γεωργία. Όλα αυτά αναφέρονται και στην έκθεση του κ. Χάτεμα. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε.